Yes, we start the meeting. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από τα σλοβενικά, τα κροατικά και τα μαλτέζικα. Μετά ε, έχουμε την έγκριση για τη δημόσια κρόση που θα γίνει στο πρώτο ήμιση του 2015 ε, εστάλει το έτοιμο αυτό σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν οι συντονιστές της Επιτροπής Απασχόλησης. Αναθεώρηση δε έχουμε τη στρατηγική της ε, Ευρώπης 2020 και το θέμα της ανεργίας και της καταπολέμησης αυτής ε, σε σχέση με τους νέους και αν είναι δυνατόν αυτό θα γίνει σε συνδυασμό και με την Επιτροπή ε, Πολιτισμού. Τρίτη ανακοίνωση. Θα έχουμε μια κοινή δημόσια κρόση για την απασχόληση και τις κοινωνικές στοιχές του TTIP το, στις Δεκεμβρίου 2014 και με την ΙΝΤΑ άλλη δημόσια κρόαση για την κατάσταση πρόοδου και ο Ιγνάσιο Γκαρσία Μπαστέρο που είναι ο βασικός μας ε, ε, διαπραγματευτής από πλευράς Ένωσης έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του. 2 Δεκεμβρίου λοιπόν οι ε, άλλες ημερομηνίες που είχαμε αναφέρει παλιότερα δεν ισχύουν. Τέταρτον, εχτες το ΔΕΚ εξέδωσε απόφαση για τη χρήση των εφαρμοστικών πράξεων στο πλαίσιο του δικτύου ε, νεότητας στο πλαίσιο, συγγνώμη, του δικτύου Γιούρες προβλέπει την εφαρμογή της πράξης Γιούρε με την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν είναι αντίθετες με τις ήδη λιμένες αποφάσεις. Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο λοιπόν και με το ΔΕΚ η Κομισιόν δεν έχει υπερβεί τις εφαρμοστικές της ε, αρμοδιότητες. Οπότε τελευταίο σημείο για αύριο είναι η Διεθνής ημέρα της εκρίζωσης της φτώχειας. Αυτό είναι απλά ενημερωτικό. Δεν θα πρέπει να μένει κανείς πίσω, να σκεφτούμε, να αποφασίσουμε και να ενεργήσουμε από κοινού και όπως γνωρίζουμε δεν έχουμε φτάσει τους στόχους τους οποίους είχαμε θεσπίσει μέσα στο πλαίσιο της Αδηγικής 2020 όσον αφορά τη φτώχεια. Η η φτώχεια αυξάνεται αντίθετα και δεν έχουμε ε, φτάσει στους στόχους μας. Ε, όμως γίνονται πράγματα στα κράτη-μέλη για την εκρίζωση, μάλλον για την εορτασμό αυτής της μέρας εκρίζωσης της στόχιας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Και μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 4. Μάλλον τελευταία ανακοίνωση αφορά τα δύο μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης στο πάνελ της ΣΤΟΑ. Έχουμε δικαίωμα σε αυτή την Επιτροπή να ορίσουμε δύο μέλη στο πάνελ της ΣΤΟΑ για τη διάρκεια 2,5 ετών. Και η συστατική συνεδρίαση της ΣΤΟΑ έχει προγραμματιστεί για τις 22 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. οι συντονιστές αποφάσισαν να προτείνουν δύο ε, ονόματα από τις δύο μεγάλες ομάδες. Το ΕΛΚ αποφάσισε να προτείνει την κυρία Γιάσλοβιέσκα και οι σοσιαλιστές τον κύριο Πεντίνσκι. Επιπλέον η η ECR έχει προτείνει την κυρία Μακιτάερ που ζητάει και το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ζητήσω ψηφοφορία να γίνει από αυτό. Αλλά αυτό που ήθελα να θίξω είναι ότι υπάρχουν 15 μέλη στο πάνελ αυτό της ΤΟΑ. Αν τους είχαμε διορίσει από το Κοινοβούλιο εν γέννη, η φυσιολογική πρακτική θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε το τύπο Ντεχόντ που θα μας είχε δώσει τέσσερις ΕΛΚ, τέσσερις σοσιαλιστές και έναν από κάθε κάθε από, μία από τις άλλες ομάδες. Όμως επειδή κάνουμε, βάζουμε δύο από κάθε επιτροπή, κάθε επιτροπή μπορεί να έχει έναν από το ΕΛΚ και έναν από το σοσιαλιστές. Οπότε περιοριζόμαστε σε αυτές τις δύο ομάδες αντί να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία και να κατανεμηθούμε με τον φυσιολογικό τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω έκκληση ότι όταν θα τελειώσουν τα μισή χρόνια να δούμε κάποια διαφορετική μέθοδο κατανομής των θέσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ωστόσο, η απόφαση των συντονιστών ήταν να ε, διοριστούν δύο μέλη από τις δύο μεγαλύτερες ομάδες. Συμφωνείτε λοιπόν να ορίσουμε τον κύριο, την κυρία Γιασλοβένκα και τον κύριο Πυρίνσκι. Μία αντίρρηση υπάρχει. Δύο. Τρεις. Ωραία, ευχαριστώ. Ελήφθη η απόφαση. Ορίζεστε λοιπόν εσείς ως μέλη ε, στο πάνελ της ΤΟΑ. Έχουμε τέσσερις ψήφους κατά. Uh, approval of minutes. No objections. Ε, Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις για την έγκριση των πρακτικών, οπότε εγκρίνονται και προχωράμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, ε, απασχόληση και κοινωνικές στοιχείες της στρατηγικής 2020. Ε, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Η Jean Lambert. Σα uh, um, Σας ευχαριστώ. Όπως θα είδατε η ομάδα μας έχει καταθέσει διάφορες τροπολογίες ε, στο ψήφισμα που συνοδεύει την προφορική ερώτηση και πρέπει απλά να σκεφτούμε κάποιες τροπολογίες για την ίδια την ε, προφορική ερώτηση. Υπάρχει ένα σύνολο τροπολογιών για την ε, προφορική ερώτηση που αλλάζει την ισορροπία του ε, ψηφίσματος θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Τώρα όσον αφορά τις τροπολογίες που ήδη καταθέσαμε στο ψήφισμα υπάρχουν διάφορες που προσπαθούν να τοποθετήσουν την διάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική διάσταση εν γέννη στη στρατηγική 2020 γιατί συχνά ακούγεται η άποψη ότι πρέπει αυτή να είναι μια συνεκτική και συνεπής στρατηγική και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία εδώ που παίζουν ρόλο και επηρεάζουν το κοινωνικό και σκέλος και το σκέλος της επασχόλησης. Πάντως θεωρούμε ότι ο τομέας που πρέπει να εξετάσει αυτή η στρατηγική δεν είναι μόνο η ίδια η φτώχεια αλλά και το θέμα της ανισότητας και της αυξανόμενης μάλιστα ανισότητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της στρατηγικής και βλέπω ότι υπάρχουν και άλλες τροπολογίες στις ίδιες γραμμές, συμβιβαστικές τροπολογίες φαντάζομαι ότι θα συνταχθούν. Ε, το πυλώνος του φίλου είναι ακόμα ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από τις πολιτικές ομάδες. Όταν βλέπουμε δηλαδή τα νούμερα που μας λένε αν προχωράμε προς τους στόχους που είχαμε θεσπίσει με την στρατηγική, δηλαδή να έχουμε ακριβή και έγκαιρη ενημέρωση, το θέμα προκύπτει και πάλι. Υπάρχει λοιπόν αυξανόμενα η άποψη ότι η επιλογή των δικτών που έχουν τα κράτη-μέλη σημαίνει πως δεν είμαστε ακόμα πλήρως σε θέση να προβούμε σε σωστή σύγκριση. Και άλλο ένα σημείο το οποίο προκύπτει από άλλα ε, κομμάτια είναι το ποιος ακριβώς ε, ασχολείται με την ανάπτυξη της στρατηγικής και βέβαια θα πρέπει να μιλήσουμε για ρόλο κλειδί των κοινωνικών εταίρων αν θεωρούμε ότι οι επιχειρηματίες είναι επίσης μέλος στρατηγικής αλλά και τα συνδικάτα ε, η κοινωνία των πολιτών όμως εδώ δεν έχει ρόλο εδώ και ενώ βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και των δεσμεύσεων έχουμε και διάφορες αναφορές στο ρόλο των κοινοβουλίων. Βλέπω πως εδώ αυτό το έχουν θέξει και άλλες πολιτικές ομάδες οπότε φαντάζομαι θα ζητηθεί ε, συμβιβαστική λύση εδώ ώστε να είμαστε βέβαιοι πως το κοινοβούλιο θα θεωρήσει πως είναι τμήμα της αξιολόγησης και της, ε, του, του απολογισμού για αυτή τη στρατηγική. Ευχαριστώ. Μπέκερ, Ελκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εμείς έχουμε μερικά σημεία που διαφωνούμε με τροπολογίες, αλλά θα συνεχίσουμε τις επαφές και τις συζητήσεις. Υπάρχουν κάποια θέματα που δεν μπορούμε να τα δεχτούμε με τη σημερινή τους εκδοχή. Για να δούμε μήπως αλλάξουν, μήπως υπάρχει δυνατότητα να τα ξαναδούμε και να προσθέσουμε και κάποια δικά μας θέματα. Κατά τα άλλα είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Ε... Ευχαριστώ. Η Γιούτα Στάιροκ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά που είπε μόλις η Τζιν Λάμπερτ μας βρίσκουν σύμφωνους σε γενικές γραμμές. Είναι πολλές ε, οι τροπολογίες που ήρθαν να εμπλουτίσουν την έκθεση. Η ε, ανισότητα, τα θέματα, τα κοινωνικά της κοινωνίας των πολιτών, ο κοινωνικός διάλογος είναι για μας ε, σημαντικά. Η καταπολέμηση της στόχιας των παιδιών κτλ. Πρέπει να μπουν και αυτά τα θέματα Οι πράσινοι έχουν κάνει πολύ καλές τροπολογίες, όπως και η και μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Κάποια προβλήματα έχουμε από την άλλη με τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των συντηρητικών ECR, γιατί για μας η άρση και κατάργηση της γραφειοκρατίας στην επιχείρηση δεν ε, θα πρέπει να σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά εις βάρος των εργαζομένων ανδρών και γυναικών. Δεν επιτρέπεται αυτό. Οπότε εκεί θα κρίνουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Ε, άλλο σημαντικό για μας, τα έχουμε ξαναπεί στην προηγούμενη συζήτηση, είναι το πίνακα επιδόσεων, το scoreboard, θα πρέπει να είναι δεσμευτικό για τα κοινωνικά για να έχουμε επιτέλους κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη και κοινωνικές επενδύσεις να εξαιρούνται από το όριο του ελλείμματος, Όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι η πολιτική λιτότητα στην Ευρώπη δεν συνοδεύεται από τη δημιουργία καλών και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Και ξέρω ότι ε, ε, ο κύριος στόχος μας είναι η πολιτική απασχόληση, αλλά και η κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να υπολείπεται και να χάνεται πίσω από τους στόχους της απασχόλησης πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και σε αυτό. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παιδική φτώχεια, επιμένω πάρα πολύ, ε, είναι πολύ σημαντικά για μας. Κατά τα άλλα, ελπίζουμε ε, στις διαπραγματεύσεις συμβαστικές που επίκυνται να έχουμε καλούς συμβιβασμούς για τον κόσμο στην Ευρώπη. Thank ευχαριστούμε, McIntyre. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ένα από αυτά που δεν μου αρέσουν είναι επειδή ε, καθοδηγούμε τις ερωτήσεις μας. Δεν ρωτάμε την άποψή τους, να μάθουμε τι πιστεύουν, ε, τους υποδεικνύουμε τι, αυτό που θέλουμε εμείς. Και η κυρία Χάρκιν και εγώ αυτό προτιμούμε. Να μην ζητάμε να συμφωνήσουμε μαζί, τους, μαζί μας, συγγνώμη, να, να ρωτάμε ποια είναι η άποψή τους. Κάποιε τροπολογίε των σοσιαλιστών δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Ε, συζητήσαμε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο ήδη. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την προφορική ερώτηση πρέπει να ε, θίξουμε αυτό το ζήτημα. για τους φραγμούς, για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ε, καλά τώρα, στο μέλλον όλα γι' αυτό θα συζητάμε, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Και για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας ε, θα γίνει συζήτηση, οπότε δεν θα σας πω τα σχετικά αυτή τη στιγμή. Θα περιμένω να γίνει σχετική συζήτηση. Ο κύριος Γκαρίκα, μπορεί μάλλον ε, να πει κάποια πράγματα γι' αυτό. Αν τώρα θέλετε στον επόμενο γύρο να ασχοληθούμε με αυτό, οκ, κανένα πρόβλημα. Ε, ευχαριστώ, Χάρκιν, από τους φιλελεύθερους. Ε, θα συμφωνήσω με την Τζίν για το θέμα της ε, ανισότητας, η αυξανόμενη ανισότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάμεσα στα κράτη-μέλη πρέπει να τονιστεί στις τροπολογίες. Ε, για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Δεν κατέθεσα τροπολογίες, όμως παρόλα αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Υπάρχει και μια άλλη τροπολογία που προέρχεται ε, και από τους πρασίνους για την επίτευξη των πέντε βασικών στόχων, συμφωνώ με αυτό. Επίσης, Υπάρχουν και αυτές οι επισφαλείς ε, προσωρινές θέσεις εργασίας και πρέπει να το αναφέρουμε. Λέω σε μια τροπολογία 40% των νέων έχουν προσωρινές συμβάσεις και 25% σε ε, ε, ημιαπασχόληση. Χρειάζεται λοιπόν αναθεώρηση της κοινωνικής κατάστασης ε, και της κατάστασης απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ένωση. Πρέπει να το συμπεριλάβουμε. Τέλος, θα αντιμετωπίσουμε και άλλη βασική δυσκολία. Τι θα συμπεριληφθεί και τι όχι στον υπολογισμό του ελλείμματος. Ίσως χρειαστεί να είμαστε ε, και ε, δημιουργικοί. Ε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί σε σχέση με τις σημερινές μας επιδόσεις. Ευχαριστώ και από την ΚΟΕ, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Ρίνια Ρονικάρη. Υπάρχει κάποιος άλλος από την ΚΟΕ. Okay. then proceed to... Όχι. Καλά, η FTD. Λαόρα Γκέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, καλημέρα. Αναλύοντας την πρόταση ψηφίσματος, λάβαμε υπόψη τις τροπολογίες που υπέβαλαν και οι συνάδελφοι μας. Ε, λυπεί ωστόσο κάπως που όταν αναφέρονται οι διάφορες ομάδες στην ανάλυση των τροπολογιών, εμείς είμαστε αγνοούμεθα. Ε, νομίζω πως ε, και εμείς δουλεύουμε για τους πολίτες μας, οπότε ίσως ε, το να λαμβάνουμε υπόψη τους συνομιλητές μας σημαίνει ότι, ότι καταφέρνουμε να συνεργαστούμε. Έχουμε υποβάλει διάφορες τροπολογίες γιατί διαπιστώσαμε ότι οι στόχοι της στρατηγικής 2020 δεν επιτυγχάνονται. Μία από τις βασικές, ένα από τα βασικά αίτια είναι ότι η απασχόληση είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται ομοιογενώς από όλε τις χώρες. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ιταλία, τη φορολόγηση της εργασίας. Εάν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε τη φορολογική πίεση στους ε, επιχειρηματίες μας που πραγματικά μπορούν να δουλέψουν ε, και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να μπορεί να μιλάμε για καινοτομία, για έρευνα αλλά ε, κύριο, πρώτο και κύριο ήταν να μειωθεί η φορολογική πίεση φτάνει στο 65% η φορολόγηση της εργασίας στη χώρα μου και στην Ευρώπη υπάρχει ανάγκη να ομοιογενοποιηθεί πραγματικά η φορολόγηση γιατί διαφορετικά για μας ε, είναι πραγματικά αδύνατο να μπορέσουμε να κάμψουμε την ανεργία και οι στόχοι που τίθεται από την στρατηγική 2020 μετά από τόσα χρόνια ε, πόρο απέχουν από την υλοποίησή τους. Οι τροπολογίες μας λοιπόν ακριβώς αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν. Τη στιγμή όπου δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης μπορούμε να βασιστούμε στην ε, καινοτομία στις νέες τεχνολογίες, ένα είδος απασχόλησης που προχωρά προς την πράσινη απασχόληση. Αυτή είναι στόχη, αλλά θα πρέπει πρώτα να, δει, να υπάρξει ένα κείμενο και να δοθεί σαφή ένδειξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ελάφρυνση προς την Ιταλία, ελάφρυνση του φόρου ε, της φορολόγησης μάλλον της απασχόλησης. Και σήμερα το πρωί ε, ο Υπουργός μάλλον ο Πρωθυπουργό είπε ότι θα μειώσει το ΙΡΑΠ, διαρκώς όμως ε, δίνει συμβουλές, καλές συμβουλές, εκεί δεν, τον, ε, ε, δεν του τη βγαίνει κανείς, αλλά συνέχεια λέει πράγματα τα οποία μετά δεν φτιάχνει. Χωρίς να μειωθεί η φορολογική πίστη του επιχειρηματίες δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο την κυρία Σαρτιέ. Ευχαριστώ. Τρία είναι τα σημεία που θέλω να σχολιάσω. Εγώ είμαι αρμόδια για το ΕΚΤ και θα ήθελα πραγματικά το... να υπερασπιστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο γιατί είναι όμοχλος ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας δεν πρέπει να συγχαίρεται με τα διαρθρωτικά ταμεία. Για θυμηθείτε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιδίωξαν να το καταργήσουν το Ευρωπαϊκό ε, Κοινωνικό Ταμείο και να το συγχωνεύσουν με το Ταμείο Συνοχής. Ε, είναι πολύ καλή ευκαιρία να τονίσουμε τη σημασία αυτού του ταμείου. Δεύτερον, ε, αυτή η πρωτοβουλία για την ε, εργασίας ε, των νέων το Συμβούλιο ασχολείται πάντοτε με τα συμφραζόμενα, με το πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται η πρωτοβουλία. Μα τα έχουμε κάνει αυτά εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε περάσει στα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα και πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί για αυτό το ζήτημα. Τρίτο σχόλιο. Βυσπαλείς θέσεις εργασίας και προσωρινές θέσεις. Μιλήσαμε για το ποσοστό των νέων σε αυτές τις θέσεις εργασίας, ε, της ε, ημιαπασχόλησης ε, και της, των προσωρινών και επισφαλών θέσεων εργασίας, θα ήθελα να προσθέσουμε εκεί και τις γυναίκες. Ευχαριστώ, Ριππέιρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ο συντονιστής του ΕΛΚ κατέθεσε μια σειρά τροπολογιών για τα ζητήματα των εξόχων απομακρυσμένων περιοχών. Όπως ξέρουμε, ε, υπάρχουν προβλήματα λόγω γεωγραφικές στήσεις, δυσκολίες στην πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες, τα δίκτυα μεταφορών, οι οικονομίες αυτών των περιοχών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και γι' αυτό ε, το ποσοστό ανεργίας ανέχει σε 24% και 51% για τους νέους. Αν ασχοληθούμε με τους μακροχρόνια δε ανέργους, βλέπουμε πόσο αρνητικές είναι οι επιδόσεις αυτό των περιοχών και έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Ένωση. Έτσι λοιπόν, ε, με βάση του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ε, κατάργηση διακριτικής ε, μεταχείρισης ε, για αυτές τις περιοχές τις απομακρυσμένε, απομακρυσμένες για να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου και να είναι ισότιμες αυτές οι περιοχές με τις λοιπές περιοχές των κρατών μελών θα πρέπει να φροντίσουμε το ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της πολιτικής 2020. Κατάλληλη πλαισίωση λοιπόν αυτών των περιοχών. Αλλιώς ισότητα με τις υπόλοιπες περιοχές δεν πρόκειται να εξασφαλιστεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ομιλήτρια από την Ιταλία μας παρουσίασε την κατάσταση στη χώρα της. Ότι είναι η φορολόγηση των επιχειρήσεων. Έχει δίκιο. Το ίδιο μπορούν να ισχυριστούν και οι Γάλλοι. Εξαιρετικά ψηλή η φορολόγηση των επιχειρήσεων. Λοιπόν, πριν κάνουμε οτιδήποτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν τη δουλειά τους για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και αν θέλουμε περισσότερα να γνωρίζουμε ο ένας για τον άλλον, θα πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ακούσαμε προηγουμένω ότι είναι κάτι άχρηστο το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Λάθος, λάθος. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο, υπάρχουν προτάσεις και μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να το ε, αλλάξουμε, να το επεξεργαστούμε. Πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν ιδέα τι εστί ευρωπαϊκό εξάμεινο. Κάποτε το αποφάσισε ως ιδέα το Συμβούλιο, καλό κτλ. Αλλά η εφαρμογή που είναι. Χρειάζεται επεξεργασία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε επί της ουσίας Έχουμε εξαιρετική τεράστια πίεση χρόνου, κάθε φορά τα ίδια. Και αν δεν τρέχουμε άρον άρον να δώσουμε μια γνωμοδότηση, μας λένε «Α, το κοινοβούλιο δεν απεφάνθη». Μα δεν είναι και το θέμα. Θα πρέπει να συμμετέχουμε ουσιαστικά και να επηρεάζουμε το περιεχόμενο. Εγώ θα επιθυμούσα ε, στο σημείο 8 ας πούμε να σκεφτούμε αυτά που λέει. 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλά, εγώ χαίρομαι για τα 6 που έχουμε ως πρώτο βήμα άλλοι αρχίζουν και πλειοδοτούν και φτάνουν και στα 21 δις και παραπάνω ε, και τα λοιπά. Τώρα το θέμα δεν είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα ή τι λεφτά θα δώσουμε σε ποιον, αλλά ποια χρήματα επενδύουμε, πού και τι αποτέλεσμα έχουν αυτά. Δηλαδή, πού υπάρχει επιτυχία και τότε μπορούμε να επιτύχουμε ακριβώς αυτούς τους κλάδους να δίνονται τα χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Όχι να αρχίζουμε να μοιράζουμε λεφτά και πού θα τα βρούμε. Σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν καν αντλήσει κονδύλια από τα έξι δις γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν οι κρατικοί μηχανισμοί και θεσμοί. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε και στις διαπραγματεύσεις. Ε, είναι σημαντικό η ε, κοινωνική πολιτική να είναι εξίσου σημαντική με ε, την οικονομική. Τι σημαίνει αυτό τώρα να ανασκοπηθούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να διεκδικήσουμε την ίση μας μεταχείριση. Υπάρχει και ευκαιρία και ο κόσμος από εμά περιμένει να κάνουμε κάτι. Thank you, Madam Κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για τους στόχους που δεν είναι δεσμευτικοί. Αυτή σε σχέση με τη μείωση της ε, φτώχειας και της ένδυας. Τα κράτη προσπαθούν να εξηγιάνουν τους προϋπολογισμούς τους. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ ε, ότι ε, η πολιτική λιτότητα σε ευθύνεται αποκλειστικά για τη φτώχεια και για τα προβλήματα και θα πρέπει να σταματήσει. Όχι. Θα πρέπει οι πόροι που έχουμε, όσο λίγοι κι αν είναι, να είναι στοχευμένοι στην επένδυσή τους η εξηγέση των προπολογισμών είναι υποχρεωτική. Έτσι κι δεν πρόκειται να αποκλίνουμε. Και ταυτόχρονα χρειάζονται κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και η δυνατότητα αντίστασης και επιβίωσης της διεθνώς είναι σημαντική. Ο Τόμας Μαν είπε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει πλήρη άγνοια για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και εγώ Τολμώ να πω ότι πρόσφατα είδα κάποια αποτελέσματα ερευνών. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ιδέα για τη στρατηγική 2020 και καλούμαστε μετά να τα εφαρμόσουμε. Αυτό με ανησυχεί βαθύτατα. Ε, είναι δική μας δουλειά αυτό. Συζητούμε με τους εκλογείς μας, με τους ψηφοφόρους, με τους πολίτες της Ευρώπης. Θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να κινητοποιηθεί και να μάθει και τι ισχύει, να διαβάσει και κανένα έγγραφο. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Thank you, Madam Chairman. Um, I... Ο κύριος Μπενιφέη. Ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για τη στρατηγική 2020 θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η καθαρή κατανομή του κονδυλίου από το πολιετές δημοσιονομικό συνιστά μείωση, καθαρά, καθαρή μείωση των ε, χρημάτων. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να υλοποιήσουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020 ε, απουσία των καταλλήλων μέσων για την εφαρμογή των μέτρων. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι να πιέσουμε για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και να ξέρουμε ποια μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για την εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής 2020. Αλλιώς θα συνεχίσουν να είναι οργισμένοι οι πολίτες εναντίον μας, ε, ε, διότι ε, πολλά υποσχόμαστε, αλλά στην πράξη δεν κάνουμε τίποτα. Ή τουλάχιστον όχι αρκετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπαν και συνάδελφοί από τους φιλελεύθερους για την ανεργία των νέων θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει με την εμπροστοβαρή εκταμείευση των 6 δις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, να εξασφαλίσουν μια χρηστή ε, χρήση των κονδυλίων και για τα χρόνια ε, εξής από το 2016 μάλλον και μετά την επόμενη προγραμματική περίοδο δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε κίνητρα. Χρειάζεται επανεκκίνηση μέσω ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής, επαναβιομηχανιοποίηση της Ευρώπης, επενδύσεις. Το είπε κάποιος και συμφωνώ. Ε, πρέπει να είμαστε ευρηματικοί για να βρούμε επενδύσεις ώστε να εφαρμόσουμε τους στόχους μας δεν θα πρέπει να μεριορίσουμε τα μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασία σε τα κράτη-μέλη. Ε, ταυτόχρονα όμως ε, θα πρέπει να μειωθεί το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα. Έχω καταθέσει και κάποιες ε, σχετικές τροπολογίες, ελπίζω να βρούμε μια συμβαστική λύση και με μια ισοσκελισμένη πρόταση να έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε την στρατηγική 2020 που προς το παρόν είναι ένα απλό ευχολόγιο δεδομένου το ότι μέσα, τα απαιτούμενα μέσα δεν τα έχουμε στη διάθεσή μας και δεν εκπληρώνουμε έτσι τις προσδοκίες των πολιτών της Ένωσης. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Θα ήθελα ξανά να θέσω το θέμα των δεσμευτικών στόχων, λέει ο κύριος Σάιμον. Δεν μας εκπλήσει αυτό. Αν οι στόχοι δεν είναι δεσμευτικοί και δεν υπάρχει νομικό καθεστώς ε, ούτε κυρώσεις για το κοινωνικό σκέλος, τότε ο κόσμος ούτε σοβαρά το παίρνει ούτε το εφαρμόζει. Στην οικονομική πτυχή υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες με ε, νομικές κυρώσεις και τα παίρνουν όλοι πολύ σοβαρά. Εμείς όσο και να μαλλιάσει η γλώσσα μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να καταστούν αυτά δεσμευτικά. Ευχαριστώ κύριε Σάιμον, διορθώνει η πρόεδρος, γιατί προ... ε, ε προφέρα ε, σου ειδικά το όνομα σας, ο κύριο Μάρτιν. Yes. Merci, Κύριος Μαρτά, ευχαριστώ Πρόεδρε ένα διαδικαστικό. Την περασμένη φορά στην Επιτροπή μας για το ψήφισμα είπατε ότι μόνο ε, οι ε, ομάδες μπορούν ε, να κάνουν τροπολογίες και μόνο στα αγγλικά. Μετά από συζήτηση δέησατε να δεχθείτε και σας ευχαριστώ γι' αυτό και οι μη εγγεγραμμένοι να κάνουν τροπολογίες και μάλιστα στη μητρική τους γλώσσα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Δυστυχώς το κείμενο το πήραμε προχτές στα αγγλικά και πρέπει να σας ομολογήσω ότι τις διάβασα ε, έτσι ακροθυγός όλες τις τροπολογίες και αυτές που έγιναν. Διαδικαστικό αυτό. Πάντως σας ευχαριστώ που μας επιτρέψατε να συνεισφέρουμε κι εμείς. των λεχθέντων, χωρίς εγώ να ξέρω πολλά αγγλικά, διάβασα τις τροπολογίες στα γρήγορα και πρώτον βλέπουμε ότι είναι σοβαρή η διαπίστωση ε, της αποτυχίας του στόχου 2020. Ε, όλοι από ό,τι φαίνεται αναγνωρίζουν ότι δεν λειτουργούν αυτά. Το βλέπουμε. Μιλάτε για την ανεργία, για τη φτώχεια, για την απασχόληση των νέων και τις θέσεις εργασίας. Αντί να αντιμετωπίσετε το κακό στη ρίζα του, όλο αυτό το δεινόν που έχουν πέσει πάνω στην Ευρώπη και και αντί να αλλάξουμε απολύτως πορεία ε, και ρότα στο 2020 έρχεται να προσθέσετε και άλλες επιβαρύνσεις και ε, προβλήματα στα κράτη-μέλη. Πουθενά δεν μιλάτε για παγκοσμιοποίηση, για ε, τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά, την οδηγία των απεσπασμένων εργαζομένων που είναι ο πραγματικός αίτιος για όλα αυτά. Εμείς κάναμε 20 τροπολογίες, αλλά από ό,τι κατάλαβα από τις συζητήσεις που είχα ε, με διάφορα μέλη που μίλησαν προηγουμένως ότι θα μας αποκλείσετε από κάθε συμβιβασμό. Μπορείτε να μας καθησυχάσετε ότι θα συμμετέχουμε τουλάχιστον στις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Every Κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να καταθέτει τροπολογίες σε οποιαδήποτε επιτροπή του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω, κάποια παρεξήγηση έγινε. Για τις μεταφράσεις τώρα. Αρχίσαμε με τα αγγλικά και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν, αν κατάλαβα καλά, τη γραμματεία. Ωραία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκύρεκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γκέρικε. Εξ ονόματος της Επιτροπής της Ομάδας ε, Συντηρητικών και Μεταρρυθμισμών σας ευχαριστώ για την έκθεση αυτή. Είναι πολύ επιτυχής. Τι είναι κοινωνικό, το έχω ξαναπεί, αυτό που δημιουργεί θέσεις εργασίας κοινωνικό, ιδιαίτερα στη στρατηγική του 2020. Η Ευρώπη θα δημιουργήσει περισσότερη εργασία εάν καταλάβει ότι η ραχοκοκαλιά μας ε, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, αν τις ενισχύσουμε θα πετύχουν διασυνοριακά. Αν έχουμε μια εσωτερική ε, αγορά για την εργασία. Μόνο τότε θα πετύχουμε. Εάν μειώσουμε τη γραφειοκρατία για τους μικρομεσαίους μας. Γενικά πιστεύω ότι από τις 166 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, πολλές έχουν και νόημα και είναι και πολύτιμες. Εμείς ως ECR τις καλωσορίζουμε. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένα που για μένα είναι ε, ευχολόγια κοινωνικής πολιτικής και δεν έχει καμιά δουλειά εδώ. Σε πολλές ε, περιπτώσεις γίνονται καλές προτάσεις για λογική ε, συμβιβαστική προσέγγιση με συμβαστικές τροπολογίες. Αν διαβάσατε τις τροπολογίες της κυρίας Μάκεντα και τις δικές μου θα διαπιστώσετε ότι θέλουμε να ληφθεί περισσότερο υπόψη ο δημογραφικός παράγων και να εστιάσουμε στις οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τρόπο θετικό. Ελπίζω να μπορούμε να προσβλέπουμε στη δική σας υποστήριξη και χαίρομαι για τις επικοδομητικές διαπραγματεύσεις που επικίνδυνται την άλλη Πέμπτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω τις ε, πρωτοβουλίες που ελήφθησαν μέχρι τώρα για την απασχόληση και ιδιαίτερα υπέρ της ε, εργασίας των νέων. Θα ήθελα όμως να τονίσω και ένα άλλο σημείο που θεωρώ σημαντικό. Η απασχόληση έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα με τις μικρομεσαίες. Για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λαμβάνουν ε, την απόφαση να προσλαμβάνουν ε, υπαλλήλους θα πρέπει να είναι αισιόδοξε για το μέλλον, να πιστεύουν στο μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε τα εξή τρία. Πρώτον, ένα σταθερό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές, να μην αλλάζει κάθε τρει και λίγο, κάθε πέντε χρόνια. Ε, ένα γενικότερο περιβάλλον ευνοϊκό. Αυτό σημαίνει και φορολογικούς κανόνες και κοινωνικές εισφορές ε, ενδεδειγμένες και προσαρμοσμένες. Το είπαν και συνάδελφοί μου προηγουμένως, αν δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Είναι πρόβλημα πραγματικό αυτό για τις επιχειρήσεις μας. Και τέλος θέλω να πω ότι η ε, απόφαση να προσλάβεις κάποιον περνάει και από μια απλούστευση των διαδικασιών μέσα στις επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν τεράστια ε, εμπόδια και διοικητικά και φορολογικά και κοινωνικών εισφορών κτλ. Λοιπόν, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας θα πρέπει να απελευθερωθεί το δυναμικό στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να είναι αυτές στην καρδιά όλου του εγχειρήματο. Ε, σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν έχω κάνει και εγώ τις τροπολογίες μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριος Κοστέλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ε, για την παράγραφο 15. Μία μικρή διευκρίνηση. Ε, καλούμε για έναν νέο κοινό δίκτυ ε, για τη φτώχεια. Εδώ καλύπτουμε δύο διαφορετικά ζητήματα, πολύ συνοπτικά και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι καλύπτεται. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ε, ότι είναι νέος δείκτης και άρα όλα τα κράτη-μέλη θα ε, χρησιμοποιούν αυτό το δείκτη και θα θυμάστε ότι η μέρος της συμφωνίας ήταν τα κράτη-μέλη ακριβώς να, ε, αν το κρίνουν ε, πρέπει να χρησιμοποιούν διαφορετικούς ε, δείκτες. Όμως αυτό δυσκολεύει την προσμέτρηση της προόδου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της στόχης κατά 20 εκατομμύρια, αν κάθε φορά χρησιμοποιούνται διαφορετικοί δείκτες σαν κράτος μέλος. Αλλά το single, το ενιαίος ε, για την φτώχεια μπορεί να ερμηνευτεί και αλλιώς. Ο δείκτης που συμφωνήθηκε σε επίπεδο ένωσης καλύπτει τρεις διαφορετικούς δείκτες, τη σχετική φτώχεια, το αναφέρουμε αυτό, ε, σοβαρή ηλική στέρηση είναι ο δεύτερος και πρέπει να λάβουμε υπόψη τη θέση των ανθρώπων στην κοινωνία και το πόσο, πόσο φτωχοί είναι σε σχέση με τους άλλους. Εάν ε, υπάρχει μια κρίση, ε, μπορεί να φαίνεται ότι μειώνεται η φτώχεια όταν ε, πλήττει τα μεσαία εισοδήματα περισσότερο από τα χαμηλά, από πλευράς δηλαδή κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό έχουμε τρεις συνιστώσεις, αν θέλετε, σε αυτόν τον ενίο δείκτη για τη φτώχεια και τυχαίνει Κάποιο τροπολογίες να το διευκρινίζουν αυτό τροποποιώντα τη διατύπωση. Θα πρέπει πραγματικά ίσω να το ξεκαθαρίσουμε ότι καλύπτονται τρία διακριτά ζητήματα μέσα σε αυτή την παράγραφο για το δίκτυο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ για όλε σας τις ε, παρεμβάσει. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει. Θα επανέλθω στους συντονιστές με διάφορες συμβιβαστικές προτάσεις εφόσον πολλές από τις τροπολογίες αφορούν παρόμοια θέματα. Θα επανέλθω λοιπόν στους συντονιστές γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα. Να σας θυμίσω επίσης για την προφορική ερώτηση ότι το πρότυπο που προβλέπετε είναι 25 σειρές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχει κανείς υπόψη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες ε, ψηφοφορίες, διότι πρέπει να ψηφίσετε. Uh, first, it's uh, the vote on the letter we will send to uh, Anderson. Λοιπόν, πρώτα έχουμε να ψηφίσουμε για την υπόθεση Άντερσεν από την Ιρλανδία ε, σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Το έχουμε ήδη συζητήσει. Ψηφίζουμε για την επιστολή χωρίς την προφορική ε, τροπολογία is it okay if we vote on the letter and the oral amendment at the same time, perhaps? Ίσως ταυτόχρονα καλύτερα την επιστολή και μαζί με την προφορική τροπολογία. Ωραία. Ψηφίστε παρακαλώ. Okay, thank you. It's carried. Ωραία. Και τώρα ψηφίζουμε για το επόμενο σημείο για την εταιρεία Sprinter της Ελλάδας, επίσης ε, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Τέλος της ψηφοφορίας. Το ΕΛΚ έχει δύο ψήφους παραπάνω. Εντάξει τώρα. Ακόμα ένας παραπάνω είστε. Ένας να βγάλει την κάρτα του. Now it's okay and it's carried. Thank you. Ωραία, λοιπόν, εγκρίνεται. Then we are on item uh, the strategic framework on health and safety at work. Um, Στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα θέματα. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπέικερ που αντικαθιστά τον κύριο Κάσα σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να περιμένω τις εξελίξεις γιατί ακόμα είμαι διάβαστος. Δεν έχω μελετήσει ε, το θέμα και με μεγάλη χαρά αφήνω την κυρία Στάιρουκ να τα πει εδώ, την παρακαθήμενη συνάδελφο. Η κυρία Στάιρουκ, ελπίζω να συνεχίσει αυτός ο ενθουσιασμός, αμύωτος για μας έρχεται πολύ αργά το πλαίσιο δράσης και είναι και πάρα πολύ ασθενές για να είμαι Και λέει θα είναι μέλος και του Refit. Αυτό μας ενοχλεί όπως και μας ενοχλούσε στο παρελθόν. Η εργασία και η, εκτός από την ασφάλεια, δηλαδή μαζί με την ασφάλεια δεν είναι γραφειοκρατικό βάρος. 4.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα και 160.000 ετησίως ε, πεθαίνουν μετά από ε, επαγγελματικές νόσους και τις συνέπειές τους. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο γραφειοκρατία αυτό για μας. Στην προφορική ερώτηση έχουμε σημαντικά αιτήματα ε, να είναι δεσμευτικά τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία και οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν, γιατί αυτοί ξέρουν ε, τα πράγματα επί τόπου, την τεχνογνωσία και να είναι σαφείς και οι ορισμοί. Ποιες είναι οι επαγγελματικές ασθένειες και ποια είναι τα εργατικά ατυχήματα. Αυτά να εγγράφονται οπωσδήποτε ως ορισμοί στο πλαίσιο. Ε, θα ήθελα επίσης να προσθέσω το εξής. οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες θα πρέπει να αποκαλύπτουν μάλλον εκείνοι που αποκαλύπτουν τις αδυναμίες και τα προβλήματα να μην μπαίνουν σε μαύρες λίστες και να στιγματίζονται. Το αντίθετο μας βοηθούν για να προχωρούμε στην Ευρώπη για τα πρότυπα ασφαλείας και θα πρέπει να προστατεύονται οι άνθρωποι αυτοί την αδιώκονται. Thank Ευχαριστώ κυρία Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να καλωσορίσω αυτή την αναθεώρηση των διαφόρων τροπολογιών περί υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας και νομίζω πως είναι απόλυτα σωστό να αξιολογήσουμε αν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκαν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σκόπιμη η αναθεώρηση τη Κομισιόν. Θέλω να καταστήσω ωστόσο σαφέ ότι ποτέ δεν πρόκειται να υποστηρίξω τη μείωση τη απαραίτητη προστασία για του εργαζόμενου. Αλλά εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό που πραγματικά πιστεύω είναι ότι αν μπορούμε να απλοποιήσουμε και να καταργήσουμε τη γραφειοκρατία, μπορούμε να αυξήσουμε το επίπεδο συμμόρφωσης. Και το λέω γιατί και εγώ η ίδια είχα μια μικρή επιχείρηση. Όταν πρέπει να περάσεις μια μέρα λοιπόν εργαζόμενος και το απόγευμα είσαι εσύ ο ίδιος ο λογιστής σου και ο δικηγόρος σου και είσαι και ο αρμόδιος για την υγεία και την ασφάλεια, πρέπει να απορροφήσεις τεράστιους όγκους, κάποιες φορές αντικρουόμενων νομοθεσιών και να προσπαθείς να βγάλεις άκρη μέσα σε όλα αυτά. Εντάξει, άμα είσαι μεγάλη επιχείρηση, έχεις τις ικανότητες να το κάνεις αυτό. Αλλά για τις μικρές επιχειρήσεις πραγματικά είναι ένας φόρτος που πιστεύω ότι εμποδίζει τις επιχειρήσεις από το να προσλάβουν περισσότερο κόσμο και τις εμποδίζει να, να έχουν ένα κάποιο βαθμό κοινή ε, λογικής. Ε, το μέσο που πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα κατά τη γνώμη μου είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερη ευελιξία στο καθορισμό του αν χρειάζονται αξιολογήσεις κινδύνου που πρέπει να καταγραφούν και να έχουν και ένα σωρό χαρτιά ε, συνοδευτικά θα πρέπει καλύτερα να δούμε το αποτέλεσμα και όχι την τεκμηρίωση. Ξέρω πως, αλλά, τουλάχιστον στο δικό μου έτσι κάνουν. Ξέρω πως άλλα κράτη-μέλη οργανώνονται διαφορετικά, αλλά εγώ θα ήθελα ε, σε όλα όσα φτιάχνουμε να απλοποιούμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την συμμόρφωση. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι υπέρ των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων. Είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου να αναπτύξουμε ένα σύστημα ε, θέσπιση στόχων και επίτευξη αυτών, πρέπει να είναι πιο στοχοθετημένε οι ενέργειε. Έχουμε μια συνήθεια και όλοι το κάνουμε του να μετατρέπουμε κάθε προφορική ερώτηση σε χριστουγεννιάτικο δέντρο και ο καθένα να βάζει το στολιδάκι του. Αλλά Ήδη είχαμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για το, για το Ναμίαντο. Ε, ε, έχουμε κάνει ένα σωρό προσπάθειες και δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Αν πραγματικά επιθυμούμε σαφή και συγκεκριμένη απάντηση από την Κομισιόν, θα πρέπει να ε, θέτουμε και σαφείς ερωτήσεις και συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και αυτό παρακαλώ να κάνει και η Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα τα πάμε καλύτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά η συνάδελφος έχει δίκιο γιατί ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από εργατικά, εργατικά ατυχήματα είναι εντυπωσιακό. 4.000 άνθρωποι κάθε χρόνο. Πρέπει να μας απασχολήσει. Πρέπει κάτι να κάνουμε και βέβαια το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε που μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Στις διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, η απάντηση σε αυτές τις ενδείξεις, ιδιαίτερα δηλαδή σε αυτή τη διαβούλευση μάλλον, κυρίως από τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες είπαν ότι ο φόρτος είναι πολύ μεγάλος για να εφαρμόσουν όλους αυτούς τους κανονισμούς. Πρέπει λοιπόν να διερευνήσουμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρξει συμμόρφωση σε ψηλού επίπεδο, αλλά ε, και πώς θα γίνει απλοποίηση εκεί όπου αυτό είναι δυνατό χρειάζονται πρακτικά και οικονομικά μέσα. Κάποιο είδος φιλικής καθοδήγησης αλλά και σωστά μέσα αξιολόγησης του κινδύνου ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, να μην χρειάζεται να επανεφευρίσκουν τον τροχό κάθε φορά να κάνουμε και κάτι, να πούμε και κάτι μάλλον για τη γύρανση του εργατικού μας δυναμικού και πώς αυτό θα επηρεάσει τις στρατηγικές για την υγεία και την ασφάλεια. Πιστεύω πως η βελτίωση των στατιστικών στοιχείων είναι σημαντική, αλλά και εδώ πρέπει πάλι να πούμε, να προσέξουμε, να μην βάλουμε υπερβολικά πολλές βαθμίδες ελέγχου και να φορτώσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, όταν το κάνουμε αυτό. Και τέλος, γιατί σε κάθε χώρο εργασία υπάρχουν οι εργαζόμενοι, υπάρχει δίκηση και αν υπάρχει κοινωνικό διάλογο, πραγματικό κοινωνικός διάλογος, ε, μπορεί αυτό με τη σειρά του να είναι ένας ε, πολύ ωραίος μηχανισμός για να εξασφαλίσουμε τη μέσα, ε, μέτρα μάλλον υγεία και ασφάλειας που να είναι πραγματικά οικονομικά. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσουμε ότι ο διάλογος είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Ευχαριστώ. Κάποιος από την ΚΟΕ θέλει να πάρει το λόγο εδώ. Όχι. Is there someone left? Κάποιος από τους πράσινους. Η κυρία Λάμπερτ έφυγε, οπότε θα πάω στο Okay, then we go to EFDD. Στην EFDD. Η κυρία Μπέγκιν, εγώ στηρίζω τις, τη θέσεις που εξέφρασαν οι προηγούμενες συνάδελφοι και εγώ θέλω να κάνω μια υπενθύμηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στην Ιταλία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι οι χωμένες μέσα σε ένα σωρό χαρτούρα που πρέπει να συμπληρώσουν καθημερινά. Όμως η ασφάλεια και στο φόρο εργασίας είναι τόσο σημαντική που δεν μπορούμε να την θεωρήσουμε μια απλή διοικητική διαδικασία ή μια ακόμα, ένα ακόμα διοικητικό φόρκο. Και εγώ το λέω αυτό πλήρη γνώση του θέματος, γιατί και εγώ είμαι πρώην ε, επιχειρηματίας και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Ε, γι' αυτό και δεχτήκαμε στην Ιταλία με μεγάλη, ε, μάλλον πολύ θετική άποψη τη νέα οδηγία για τις συνθήκες εργασίας και για έναν επιπλέον ε, ασφάλιση. Και εγώ θα πρέπει να σας πω ότι ε, άνοιξα ένα κομμάτι, ένα παράρτημα ε, στην εταιρεία μου για να καλύψω αυτό το θέμα και το, μετά το έκλεισα γιατί στην Ιταλία ποτέ δεν, δεν λειτουργήσε. Στην Ιταλία καταφέρνουν με μερικά ευρώ να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια online και να τελειώνει υπόθεση. Η στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το στρες είναι πιο πολύ από ό,τι στις μεγάλες γιατί υπάρχει πραγματική δυσκολία για έναν εργοζόμενο να καταγγείλει δύσκολες καταστάσεις. Πραγματικά λοιπόν πρέπει να βρούμε ένα σημείο επαφής ανάμεσα σε αυτό που είναι οι δίκαιες απαιτήσει των μικρών επιχειρηματιών που πρέπει να φτάσουν το τέλος του μήνα και να δημιουργήσουν νέα απασχόληση, νέα απασχόληση και τη θεμετή επιθυμία ε, οποιοδήποτε να ζει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον και που του επιτρέπει να αναπτύξει όλο του το δυναμικό. Δυστυχώς οι επιχειρηματίες δεν καταλαβαίνουν ακόμα ότι όταν ένας άνθρωπος εργάζεται νυφάλια στο χώρο εργασία τους παράγει πολύ περισσότερο. Simon, Ευχαριστώ. Σάιμον. Σας ευχαριστώ. Για το θέμα της μείωσης του φόρτου στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όλοι θέλουν να μειώσουν τη γραφειοκρατία όταν αυτή περιτεύει. Αυτό είναι βέβαιο και ίσως να μην χρειάζεται να συμπληρώνουν τις ίδια, τα ίδια έντυπα μια, οι μεγάλες επιχειρήσεις με μια οικογενειακή επιχείρηση. Ωστόσο, τα δικαιώματα και η υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων, είτε στη μία είτε στην άλλη επιχείρηση, πρέπει να προστατεύονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Και όταν μιλούμε σε εκπροσώπους των μικρών επιχειρήσεων λένε, το λένε αυτό ξεκάθαρα. Εμείς αναμένουμε να έχουμε την ίδια ακριβώς ε, απόδοση από τους μικρούς εργοδότες όπως και από τους μεγάλους. Αλλά αυτό δεν γίνεται πάντα σαφές στα λόγια των δεξιών ομάδων εδώ όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να καταστεί απόλυτα σαφές, να είναι καταγεγραμμένο, να μην υπάρχει καμιά αμφισημία απολύτως, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικών ειδών δικαιώματα, και να προστατεύεται μερικώς η υγεία κάποιων. Όχι, πρέπει να είναι παντού ακριβώς τα ίδια, ενώ θα μειώνεται το γραφειοκρατικό βάρος όπου αυτό είναι δυνατόν. Η κυρία Μάκινταρ είπε, ρώτησε γιατί να χρειάζεται να επανέλθουμε στον αμύαντο και είχαμε και εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας κτλ. Μα αυτό εδώ υποτίθεται ότι είναι στρατηγική. Υποτίθεται ότι είναι κάτι το οποίο καλύπτει ε, όλες τις ε, πτυχές ε, για πολλά χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός κάτι που είναι τόσο σημαντικό και που εξακολουθεί να σκοτώνει χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο. Γιατί να το αφήσουμε από εκτός. Αφού είναι σημαντικό πρέπει να είναι μέσα στην πιστατική. Και Αφού χιλιάδες κόσμος συνεχίζει να πεθαίνει από αυτό, πρέπει να συνεχίσουμε και εμείς να το λέμε. Να λέμε να υπάρχει μητρό για τον αμύαντο, να υπάρχει μεγάλη κατάρτιση, πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν και αν εμείς δεν το, δεν το αναφέρουμε και δεν το ρητά και ξεκάθαρα, τότε ποιος θα το κάνει. Το ίδιο για τα, τις καρκινογόνες ε, ουσίες. Πού πήγε γι' αυτό. Και τέλος, για τις μικρές επιχειρήσεις. Να μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, στον τομέα των κατασκευαστικών, όπου τα θέματα υγείας και ασφάλειας είναι τεράστια σημασία, όπου και πάλι χιλιάδες κόσμος σκοτώνεται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν ε, κάποιες, κάποιοι τεράστιοι, πάρα πολύ πλούσιοι, πολυεθνικοί παίκτες στην κατασκευαστικό τομέα, όπου σχεδόν όμως κανένας εργαζόμενος δεν απασχολείται άμεσα από αυτούς τους τεράστιους εργοδότες, αλλά από υπεργολάβους που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ήταν τελείως λάθος αν αυτοί οι υπεργολάβοι και οι εργαζόμενοι που αυτοί προσλαμβάνουν θεωρηθούν εργαζόμενοι μικρών επιχειρήσεων, ενώ στην ουσία είναι εργαζόμενοι για τεράστιες πολυεθνικές που κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ κάθε χρόνο. Simon, Ευχαριστώ. Ο Ρολάν. Ρολάν, ευχαριστώ, από την προσωπική μου επαγγελματική εμπειρία έχω ζήσει πολλά εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες σε μια σειρά από κλάδους. Έχω να πω λοιπόν τα εξή ζητήματα. Πρώτον, η στρατηγική που έχουμε είναι όντως πολύ αργή στην υλοποίησή της και επίγει πάρα πολύ. Για τους εξή δύο λόγους. Και το ανθρώπινο στοιχείο προφανώς, το ακούσαμε 4.000 ε, νεκροί το χρόνο, 3 εκατομμύρια σοβαρά ατυχήματα και δεν μιλώ για τις αναπηρίες που απορρέουν από εργατικά ατυχήματα. Αυτό έχει και οικονομικό κόστος πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή βαραίνει και τη ζωή των επιχειρήσεων ε, και τους κρατικούς προϋπολογισμούς πάρα πολύ, δηλαδή μέσω της κοινωνικής ασφάλισης. Ε, πέφτουν λίγο οι στατιστικές και μας χαροποιεί αυτό, αλλά αλλάζουν και οι συνθήκες εργασίας και αλλάζουν και τα εργατικά ατυχήματα, εξελίσσονται τα επαγγέλματα. Όταν είναι λιγότερο χειρονακτικά και πιο πνευματικά τα επαγγέλματα είναι και λιγότερα τα ε, ατυχήματα, τα σωματικά, αλλά είναι νέες ασθένειες που εμφανίζονται, όπως είναι υπερκόπωση, burnout και θα μπορούσε να ακολουθήσει μακρύς κατάλογος στα θέματα αυτά. Επίσης και στα προϊόντα, αλλάζουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Άρα όλα αυτά χρειάζονται παρακολούθηση, εναρμόνιση. εκπλήσουμε αρκετά βλέποντας την κατάσταση από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν ορισμένα προϊόντα που σε κάποια χώρα θεωρούνται καρκινογόνα και επειδή περνά στα σύνορα λίγο χιλιόμετρα παρακάτω είναι εντάξει. Κανένα πρόβλημα για τους γείτονες που το χρησιμοποιούν. Ε, ε, ε, είναι τέσσερις οι λέξεις κλειδιά για να προχωρήσουμε σε αυτή την ιστορία και να μειωθούν τα ατυχήματα, οι νεκροί και οι άρρωστοι. Είναι η πρόληψη πρώτον. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, η ενημέρωση η διαβούλευση με κοινωνικό διάλογο και ο έλεγχος. Αυτά τα τέσσερα. Και όταν μιλώ για έλεγχο, εννοώ τα εξή δύο. Έλεγχος για να γίνεται σεβαστή η νομοθεσία και οι κανονισμοί, αλλά και ιδίω για τι μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος υπό μορφή πληροφορίας και καθοδήγηση. Πόσε φορέ δεν έχω συναντήσει εταιρείε που ε, παραλίγο να πτωχεύσουν γιατί δεν εφήρμοζαν μια ε, νομοθεσία που δεν είχαν καταλάβει. Ε, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι προστασίες για τους εργαζομένους και υπήρξε ένα θανατηφόρο ατύχημα, δεν ε, το κάλυψε η ασφάλεια γιατί δεν τηρήθηκαν οι κανόνες και είχε τεράστιες δυσκολίες οικονομικές επιχείρησεις. Η απλούστευση. Όλοι μπορούμε να συμφωνούμε ότι είναι ανάγκη να απλουστευτεί η νομοθεσία και να ελαφρυνθεί. Αυτό δεν γίνεται ποτέ όμως ε, θέτοντας σε κινδύνο την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα, τα στατιστικά στοιχεία πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα για τα θέματα της ασφάλειας στην εργασία. Ε, θα μιλήσω για τη χώρα μου, γιατί πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς καν να είναι ασφαλισμένοι. Οπότε όταν του συμβεί κάποιο ατύχημα στην εργασία δεν θεωρείται καν εργατικό ατύχημα. Λοιπόν, Πρωταρχικό μέλημα φαντάζομαι θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν ασφάλεια και να υπάρχουν όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την προστασία τους στην εργασία. Ευχαριστώ. Thank you. You might also add that small Ευχαριστώ. Μπορείτε να προσθέσετε ότι μικρές, για τις μικρές επιχειρήσεις όταν συμβεί κάτι με τους εργαζομένους αυτό μπορεί να είναι καταστροφή και για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι μεγάλες έχουν ασφάλειες, έχουν ε, πολύ προσωπικό. Άρα για τις μικρές επιχειρήσεις ε, είναι καλό να ισχύσουν αυστηρότεροι κανονισμοί. Για να ακούσουμε την Επιτροπή. Ο κύριος Λεγκάλ. Uh, Ευχαριστώ. Δεν έχουμε σχόλια. Ε, υποβάλλετε εσείς μια προφορική ερώτηση, θα απαντήσουμε στην Ολομέλεια. I lost you. Miss, Miss Regner. Δεν σας είδα κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, όταν κάθεται κανείς σε αυτή την ωραία αριστερή γωνιά, συχνά τον παραβλέπει το Προεδρείο. Ε, Θέλω να συμπληρώσω μερικά πράγματα. Ωραία. Πρόληψη, ενημέρωση, κοινωνικός διάλογος. Τεράστια σημασία όταν σκεφτόμαστε τη στρατηγική μας. Θέλω όμως πολύ απλά να τα ξαναπώ. Όταν μιλούμε για υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν πρόκειται ε, για ε, το κερασάκι στην τούρτα, αλλά για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι τόσο σημαντικό, ώστε σε αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να το έχουμε πάντα γνώμονα και οδηγό μας. Το θέμα δεν είναι ε, η άρση της γραφειοκρατίας να έχει ως τίμημα την ασφάλεια και την υγιεινή συνεργασία δεν είναι το ένα ή το άλλο, όλα σημαντικά και στις μεγάλες και στις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να είναι ο φάρος μας ε, σε αυτή την εργασία και η επεξίδα. Και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που έχουμε να κοιτάξουμε δεν είναι μόνο πιο πνευματικά τα επαγγέλματα και λιγότερο χειρονακτικά αλλά όλο και πιο πολύ βλέπουμε κάτι που δεν θα το είχαμε καν σκεφτεί πριν από μερικά χρόνια. Ε, μικρά ε, μαγαζιά ε, σε υπόγειους σταθμούς του μετρό. Τι κάνουν οι εργαζόμενοι που είναι όλη μέρα στο σκοτάδι και σε αυτή τη ζέστη ή στο σούπερ μάρκετ όταν δουλεύει κάνος όλη, όλη μέρα μπροστά στα ψυγεία. όλα αυτά είναι νέα ζητήματα που πρέπει να κοιτάξουμε. Γνωρίζετε όλοι το παράδειγμα αυτό, αλλά καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε συχνά. Αυτή η συμφωνία για τους κομμωτές και τους κουρίς. Ε, αυτό είναι εύγλωτο και μιλάει για πολλά άλλα επαγγέλματα. Θέλω να πω στην κυρία Μακιντάιερ το εξής. Αυτό έχει να κάνει και με τους εργοδότες. Ε, οι ε, ε, κομμωτές είναι μικρά κομμωτήρια και από την Αγγλία και από αλλού που λέγουν ότι αν βάλουμε γάντια, όπως έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί εταίροι, αυτό δεν σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία, είναι περισσότερη ασφάλεια. Όταν μπαίνει στα μάξια, αμέσω βάζει τη ζώνη ασφαλείας. Αυτόματα, εγώ θα πρέπει να βάζω γάντια. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να συνεννοούμαστε πάντα και να ρωτούμε και εκείνους που ξέρουν τα πράγματα καλύτερα, οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες, ας τους ακούμε αυτούς, ας τους αφήνουμε να πούν τη γνώμη τους και να μην παρουσιάζουμε απλουστευτικά τα αποτελέσματα και να δείχνουμε μόνο τα αρνητικά, όπως είναι στο Refit. Λιγότερος λαϊκισμός χρειάζεται και περισσότερη προσοχή. Είναι θεμελιώδη αυτά τα δικαιώματα. Thank uh, ευχαριστούμε, κυρία Ρέγνερ. Κύριο Κρασεντεύσκη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω ένα ζήτημα μόνο. Είπανε πολύ ότι ότι είναι περίπλοκα τα μέτρα και δύσκολη εφαρμογή τους σε μικρές και μισές επιχειρήσεις. Η κοινωνική πραγματικότητα όμως μας δείχνει πως ε, αυτοί οι περίπλοκοι κανόνες, εγώ δεν έχω προσωπικά επιχείρηση, αλλά γνωρίζω τους κανόνες ε, με την ιδιότητα του εργαζόμενου. και πιστεύω ότι ε, ο εργαζόμενος δεν έχει κανένα πρόβλημα να προσυμφέρουν προς συμφέρον αυτοί οι αυστηροί κανόνες. Εγώ προέρχομαι από την αποκαλούμενη κεντρική και ανατολική Ευρώπη και ξέρω ότι ε, όταν είναι υπερβολικά περίπλοκα τα μέτρα και αδυνατούν οι επιχειρήσεις ε, να τα εφαρμόσουν, τότε απλώς αγνοούνται και το ίδιο προτείνεται και στους εργαζομένους. Αγνοήστε τους κανόνες, τους λένε. Ε, και παραδείγματος χάρη υπάρχει παραγνώριση των κανόνων και μη καταβολή αποζημιώσεων παραδείγματος χάρη. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα, να απλουστεύσουμε τους κανόνες, ώστε να λειτουργούν προς συμφέρον των εργαζομένων. Νομίζω ότι απέχουμε λίγο από την πραγματικότητα. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη κανόνων ε, στα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα είναι ότι αγνοούν οι επιχειρήσεις τους κανόνες. Για τις αναρωτικές ε, άδειες, ε, παραδείγματος χάρη, συχνά αγνοούνται οι κανόνες και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν εξυπηρετούνται ούτε το συμφέρον ούτε της επιχείρησης ούτε του εργαζομένου. Χρειαζόμαστε απλούστερους κανόνες. Γιώτα Στάινμπρουκ. Λοιπόν, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κομισιόν, Συμβούλιο, Πολιτική δεν θα πρέπει να ισχυριζόμαστε, να έχουμε αυτή την αλαζονία, ότι γνωρίζουμε ή ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από τους κοινωνικούς εταίρους που είναι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Αυτοί ξέρουν την κατάσταση επιτόπου, ξέρουν τι ανάγκες έχουν για την ε, προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας. Η Εύλεν Ρέγνερ το είπε, είναι θεμελιώδη δικαιώματα αυτά. Όταν υπάρχουν συμφωνίες τι δουλειά έχει η πολιτική. Δεν χρειάζεται να τις ελέγχει και να τις δοκιμάζει αυτές τις συμφωνίες. Να ακούσουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα που έχουν εργαστεί στην εκπόνησή τους. Δεν είναι τόσο περίπλοκο πολύ συχνά. Είναι συχνά πολύ ακριβό για κάποιους. Το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Ε, ποιο είναι το κόστος για την κοινωνία μετά. Αν τα καταργήσουμε αυτά. Το κοινωνικό σύνολο έρχεται να τα πληρώσει. Εντάξει, εξοικονομούν λεφτά κάποιες εταιρείες και μετά πληρώνει την ύφη η κοινωνία ολόκληρη και πολύ πιο ακριβά. Όταν υπάρχουν τέτοιες κοινωνικές συμφωνίες δεν θα πρέπει να τις καταργούμε με σύνθημα η επικεφαλίδα κατάργηση ε, γραφειοκρατίας. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς εταίρους όταν συμφωνούν και ε, καταλήγουν και το λέω και εξ ονόματος της ομάδας μου, θα πρέπει η πολιτική να κάνει ένα βήμα πίσω και να πει αυτοί τα ξέρουν καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ο κ. Δομινίκ Μαχτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να συμφωνήσω με τη συνάδελφο. Για να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία. Ε, είναι εφαρμόζονται καλά οι κανόνες, προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό οι εργαζόμενοι, όμως ε, στα ε, ναυπηγεία ή στα δημόσια έργα ή ε, οικοδομικές εταιρείες χρησιμοποιούν αποσπασμένους εργαζόμενους που υπάγονται στους κανόνες της χώρας προέλευσης. Τι σημαίνει αυτό, χρειάζεται εναρμόνιση, όχι τόσο όχι υπερβολικά περιοριστικοί κανόνες γιατί δεν εφαρμόζονται όπως σωστά επί συναδελφός, να βρούμε μια μέση λογική λύση ούτω ώστε να ε, καταργήσουμε αυτή την ανισότητα. Σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προστατεύονται παρκώς ε, οι εργαζόμενοι. Σας ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις, λέει η κυρία Ούλσκοκ. Έγινε η πρώτη λοιπόν ανταλλαγή απόψεων. Στην δεύτερη ε, σύνοδο του Νοεμβρίου θα υποβάλω αυτή την προφορική ερώτηση. Απευθυνθείτε παρακαλώ συντονιστές ε, για να προσθέσετε σχόλια. Θα περνάτε κάθε φορά από τον συντονιστή της πολιτικής σας ομάδας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στις 12. Αυτή είναι καταληκτική προθεσμία για περαιτέρω σχόλια. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα περάσουμε στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων για την προφορική ερώτηση για την ε, εφαρμογή της οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία. Το στείλαμε ε, στις 13 Οκτωβρίου σε όλους το κείμενο βασίζεται στην ε, κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας ε, για την εφηλετική ισότητα και την οδηγία για την ισότητα ε, στην απασχόληση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπέκερ. Äh, Εμεί στην ομάδα μας δεν διαφωνούμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση με το έγγραφο που έχει κατατεθεί, οπότε θα περιοριστώ σε αυτή τη θετική αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στάινροκ. Και εμεί θεωρούμε ότι το πρώτο σχέδιο είναι καλό και πολύ καλό μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικές οι οδηγίες αυτές που θα πρέπει επιγόντως να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία, στα κράτη-μέλη. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμένα είναι να εφαρμόζονται καλύτερα και να υλοποιούνται. Και οι άνθρωποι να γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν επί τόπου, ιδιαίτερα στην οδηγία για την ίση μεταχείριση, στην απασχόληση και στα επάγγελματα. Εμείς ως Επιτροπή, λέω, κοινοβουλευτική, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι και να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία αυτή την οδηγία. Είναι το σημαντικότερο όλων στη δουλειά μας. Well, thank you for... Σας ευχαριστώ Τα ίδια με την προηγούμενη προφορική ερώτηση. Α, οι υπόλοιποι συντονιστές μου στέλνουν το λόγο. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ πολύ σύντομη θα είμαι πρόεδρε. Ε, και εμείς υποστηρίζουμε το περιεχόμενο της προφορικής ερώτησης. Κάποιες ίσως σημασίες αλλαγές ίσως να επιφέρουμε. Ε, εκεί που λέει για την έλλειψη ευαισθητοποίησης ε, λόγω του σοβαρού προβλήματος της μη υποβολής εκθέσεων και στοιχείων είναι σημαντικό να το αναφέρουμε για τη συντολογή δεδομένων υπάρχουν ε, κάποια, κάποιες ανησυχίες για το άχθος που συνεπάγεται αυτή η συλλογή δεδομένων και θα χρειαστεί να το συζητήσουμε. Από ό,τι βλέπω, αν ερμηνεύω σωστά την έκθεση της Επιτροπής, είναι απαραίτητα τα καλά δεδομένα για να εξασφαλίσουμε βέλτιστες πρακτικές ε, στα κράτη-μέλη, κυρίως ε, για τις περιπτώσεις ε, έμεσης και πολλαπλής διακριτικής μεταχείρισης. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Εν γέννη πάντως θα υποστηρίξουμε σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο αυτής της προφορικής ερώτησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Η κυρία Στίβενς από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ κυρία Στέβενς, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα και εγώ εξ ονόματος της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών να υποστηρίξω πλήρως αυτή την προφορική ερώτηση. Αλλά όπως ε, είπε και η προλαλή σας, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που πρέπει να κάνουμε. Και βέβαια περιμένουμε και εμείς από όλες τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας ε, επιτρέπουν να είμαστε εγκαίρως ενήμεροι για να μπορούμε να ε, δρούμε και να αντιμετωπίζουμε κάποιες παρενέργειες και κάποια ανητικά και για τις δύο οδηγίες. Λοιπόν, παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο συγκεκριμένη στα όσα λέγει και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε και μια συγκεκριμένη απάντηση όταν είναι όλα γενικά και αόριστα την απαντήσεις ε, και έχω τις εξής προτάσεις πρώτον να Τι σημαίνει καλύτερη εφαρμογή στην πράξη και υλοποίηση. Πολύ λόγια του αέρα είναι αυτά, οριστολογίες και ευρύτατο το πεδίο. Θα πρέπει πιο συγκεκριμένα να τα λέμε και να ε, κάνουμε προτάσεις. Θα το πω και στους συντονιστές αυτό. Και μια δεύτερη ερώτηση. Τι θα πει έλλειψη συνειδητοποίησης. Χαιρετίσματα. Και αυτό είναι ευρύτατο τι είναι αυτό, ότι δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε δεδομένα, δεν έχουμε πληροφορίες. Θα πρέπει να είμαστε πιο χειροπιαστοί, πιο συγκεκριμένοι. Να το εξηγούμε, να, το κατονομάζουμε. Τι είναι αυτή η διαχείριση, ρατσισμός για άτομα με ξένη προέλευση, με αναπηρία, τι θα, γενικά μιλάμε για διακρίσεις, να πούμε με το όνομά τους ποια είναι αυτά αν είναι η αναπηρία, είναι η θρησκεία, είναι η καταγωγή. Θέλω πιο συγκεκριμένη κατανομή και επιμερισμό. Υπάρχει και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει κυρώσει αυτή και στη σύμβαση της, το ΓΟΙΕ λέει ότι διάκριση είναι όταν δεν υπάρχει ε, η σωστή μέρημνα για προσαρμογή του χώρου εργασίας στο άτομο με αναπηρία. Για την πρόσβασή του δηλαδή. Ε, λέτε γενικά και αόριστα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτό πολύ συχνά στην πράξη δεν θεωρείται ότι συνιστά διάκριση. Τι έχει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει συμπεριληφθεί η σύμβαση του ΟΗΕ στην οδηγία ή όχι. Θα τα πω και στο συντονιστή μας, αλλά ήθελα να τα πω και εδώ. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, is there some... Σας ευχαριστούμε. Εκπροσωπεί κάποιος την Κουέμπος, ήρθε κάποιος στο μεταξύ. Uh, from the... Από τους πράσινους. Ούτε. Η FTD. Εσείς ίσως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι και εμείς στην ομάδα μας θα στηρίξουμε το αίτημα για προφορική ε, ερώτηση. Θα το συζητήσουμε και εσωτερικά βέβαια, αλλά και εγώ είμαι υπέρ της μεγαλύτερης ε, ε, συνέπειας και πιο, του πιο συγκεκριμένου, σε πιο συγκεκριμένη σύνταξη. Ευχαριστώ, Μαρτά. Merci, Madame le Président. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίω τα όσα άκουσα είναι αξιέπαινα. Κατά πολέμηση του ρατσισμού όλοι εδώ είναι υπέρ. Όμως εγώ θα ήθελα να ε, πιστήσω την προσοχή της Κομισιόν σε αυτό το σύστημα θετικής, ε, θετικών διακρίσεων το οποίο μπορεί να φτάσει στα άκρα και ε, φοβάμαι και γι' αυτό θέλω να σας προειδοποιήσω ότι μέσα σε ένα κλίμα επισφάλειας και που ισχύει σε όλες τις χώρες μέλη αυτή τη στιγμή, αυτή η θετική διάκριση μπορεί να ερμηνευτεί ως ε, μια προτίμηση στους ε, αλλοδαπούς. Προσέχετε λοιπόν τι λέτε, γιατί αυτή η προσωμείωση στην προτίμηση σε αλλοδαπούς για τον κόσμο που είναι σε επισφάλεια στη χώρα του θα αυξήσει τις ρογμές ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες. Προσοχή μεγάλη λοιπόν. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είστε την κυρία Λίντχορ. Uh, Η Κομισιόν καταγράφει όλα όσα υπόθηκαν και θα προετοιμάσουμε την απάντηση μας ε, αναλόγως. Απλά θα ήθελα να γνωρίζω σε σχέση με το σημείο της λογικής ε, ε, πρόβλεψης για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό ήδη είναι εγγυημένο μέσα στις σχετικές οδηγίες. Δεν είναι μόνο στη σύμβαση αλλά και στην οδηγία. Και όσον αφορά τη θετική διάκριση Οι οδηγίες επιτρέπουν στα κάτι μελη να αναλάβουν θετική δράση εξ των ανθρώπων με... που, υφίστανται διακρίσεις, αλλά δεν τα υποχρεώνει να κάνουν συγκεκριτικές δράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευκρινήσεις σας και τώρα θα προχωρήσουμε. στην έγκριση στην Επιτροπή Επασχόλησης 4 Νοεμβρίου και η προφορική ερώτηση θα κατατεθεί από εμένα εξ ονόματος Επιτροπής γιατί στη δεύτερη σύνοδο του Νοεμβρίου. Στο όνομα των Προέδρων, ε, λοιπόν, ε, θα υποβληθεί η προφορική ερώτηση για τη δεύτερη σύνοδο. Σας ευχαριστώ πολύ και η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 4 Νοεμβρίου. Έχουμε κάνει όλα όσα έπρεπε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας.